έχω και άλλες ε, θλιβερές ανακοινώσεις. Στις 19 Δεκεμβρίου ε, πέθανε ο συνάδελφος Φιλίπ Πρέτμπορν 63 ετών κατόπιν βαριάς ασθένειας. Ο συνάδελφος Πρέτμπορν ε, ήταν από το 96 βουλευτής εδώ και όποιος τον γνωρίζει, το εκπροσωπούσε ε, με μεγάλη περηφάνεια την περιοχή του, το West Midlands. Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία ε, ως πολεοδόμος. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, εξέφρασα ήδη τα θερμά μου συλλημητήρια και θα ήθελα ε, να το επαναλάβω εδώ, δεν θα τον λησμονήσουμε. Στις 26 ε, Δεκεμβρίου του περασμένου έτους πέθανε ο Λέο Τίντεμαντς σε ηλικία 92 ετών ε, στο σπίτι του κοντά στην Αμβέρσα, ο οποίος ήταν βαθιά επηρεασμένος από τη βάναυση κατοχή της χώρας του από τους Ναζί, οι οποίοι όταν ήταν 18 ετών τον ανάγκασαν στην φυγή. Αλλά ο Τίντεμαν ολόκληρη τη ζωή του εργάστηκε για την υπόθεση ειρήνης στην Ευρώπη. Ως βουλευτή του Βελγικού Κοινοβουλίου, ως ε, Πρωθυπουργό ε, του Βασιλείου του Βελγίου, ως υπουργό εξωτερικών της χώρας του και ως ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι πρώτε άμεσε εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Τίντεμαν εξελέγει στο Βέλγιο με τέτοια πλειοψηφία που οι εφημερίδες τότε τον αποκάλεσαν Mr. Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι πραγματικά ο τίτλος αυτός του ταιριάζει γιατί ασφαλώς υπήρξε ένας μεγάλος ευρωπαϊστής. Ε, προς την οικογένειά του, εξ ονόματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μας ε, συλληπιτήρια. Πραγματικά θα τον κρατήσουμε ζωντανό στη μνήμη μας και παρακαλώ για να τιμήσουμε τους δύο συναδέλφους να σηκωθείτε.